συνάδελφοι και καλώς ορίσατε μετά τις διακοπές, μετά το διάλειμμα αυτό. Εγκρίνετε παρακαλώ η μερίστη διάταξη. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2017. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ε, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Αύριο θα κάνω τις ανακοινώσεις του Προέδρου σε ό,τι αφορά και τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις και ας περάσουμε πάρα αυτό στο σημείο 6 της σημερινής συνδιαταξής για το FinTech την έκθεση για την FinTech όπου και καλούμαστε να εξετάσουμε τις τροπολογίες είναι εδώ και η Κόρα Πανιουνχάιζεν, η συγκεκριά μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η FinTech θα είναι η καινούργια αλλάξη της μόδας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυτό μάλιστα με εδώ κάποιο καιρό και στη ΣΥΠΑ και στην Ασία άλλωστε. Στην Ευρώπη μόλις ξεκινούμε να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της FinTech σε διάφορα συνέδρια. Ε, ρωτάω διάφορους φορείς ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των bitcoin και συνήθως κανένας δεν σηκώνει το χέρι του. Και αυτό θεωρώ σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για το μέλλον. Άρα, στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε κατά νου φυσικά κατά πόσον ε, θα μας χτυπήσει άλλη κρίση. Αλλά να έχουμε και υπόψη μας τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί αν δεν παρακολουθήσουμε την όλη λογική του FinTech, ε, δεν θα είμαστε σε ηγετική θέση. Πιο πολλέ επενδύσει ω τώρα έχουν γίνει στην Κίνα, στη ΣΥΠΑ, στο Ισραήλ και γι' αυτό λοιπόν οι πιο πολλέ εταιρείε FinTech εκεί ακριβώ βρίσκονται. Και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική ακόμα έχει καλύτερη προβάδισμα η FinTech. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ανταγωνιστική και να έχει την υποδομή, την εξαιρετική αυτή που έχει, θα πρέπει αυτά να γίνουν κανόνα και όχι εξαίρεση. Και αυτό και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Η FinTech οδηγεί σε πιο πολύ διαφάνεια, μεγαλύτερες επιλογές, καλύτερες ε, υπηρεσίες, καλύτερο και χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. Και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος μπορεί να υποφεληθεί από εξελίξεις FinTech όπως είναι το Big Robot και ε, Big Data και το Robot. Επίσης, καλύτερη διαχείριση κινδύνου συνεπάγεται η FinTech. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη της FinTech θα πρέπει να διευκολυνθεί και όχι να καταπατηθεί και να περιοριστεί η επιρροή της FinTech. Συνολικά λοιπόν συνάδελφοι θέλουμε να βελτιώσουμε το κείμενο της έκθεσής μου και πολύ χαίρομαι που δεν θα συζητήσουμε, μάλλον δεν μπορούμε να συζητήσουμε στη συνεδρίαση αυτή όλα τα τεχνικά στοιχεία, αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον φτάσαμε σε μια πολιτική συμφωνία και έχουμε κοινέ προτεραιότητε, εν πάση περιπτώσει. Και η πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Ο εικονικό ε, ληστή, ο οποίο μπαίνει μάλλον σε μια τράπεζα και με το όπλο του κραδένει και απειλεί του υπαλλήλου, ε, υπάρχει μόνο στι ταινίε πλέον. Σήμερα είναι hacker αυτό και λειτουργεί από την αποθήκη του. Η ασφάλεια είναι αυξανόμενο πρόβλημα παγκοσμίω και σύμφωνα με την Κανθόρτα το έγκλημα κοστίζει 200 δισεκατομμύρια ανά έτο σε παγκοσμίο επίπεδο. Ενώ με άλλε εκτιμήσει, ε, η οικονομική ζημία για την κοινωνία κινείται πιο πολύ στα 400 δις ε, ευρώ. Συγγνώμη, δολάρια. Και σήμερα είδαμε σε ένα ρεπορτάζ ότι στη Γερμανία πέρσι ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων διπλασιάστηκε. Νομίζω ότι λοιπόν αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Και πάνω από 80% των ψηφιακών δεδομένων ε, στον κόσμο δεν έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό καταδεικνύει πόσο εκθετικά έχουν αυξηθεί οι ροές δεδομένων τα τελευταία χρόνια χρόνια. Αυτό αποτελεί μεγάλη πηγή ανησυχία. Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε καλύτερα στην ασφάλεια, στι τράπεζε, σε άλλα χρηματοπιστικά ιδρύματα και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα στρέστ. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει σωστή ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών μεταξύ εταιριών και κυβερνήσεων, γιατί είναι μεγάλο το διακύβευμα και για του επιχειρηματίε και για τι κυβερνήσει και για του καταναλωτέ. Ο μελλοντικό ε, χρηματοπιστωτικό ε, κλάδο θα χρειάζεται πιο πολύ τεχνικό προσωπικό, όχι τόσο πολύ δικηγόρου κτλ. Όχι μόνο για την δημιουργία αλγορίθμων, αλλά και για την προστασία των τεράστιων ροών δεδομένων. Και το ίδιο ισχύει και για του χρηματοπιστωτικού ε, ρυθμιστές. Θα πρέπει να καταλαβήσουν την περίπλοκη δομή των εξέλιξεων fintech για να κατανοήσουμε πως η fintech χρειάζεται και συνδέεται με την πραγματική οικονομία πρωτού λαμβάνουν αποφάσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχουν νέοι φορείς οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά fintech και η fintech δεν είναι μόνο για τις παραδοσιακές τράπεζες και τους ασφαλιστές, αλλά και πολλοί, πολλές startups βρίσκονται και αναμειγνύονται στην fintech και η Apple, Apple Pay, Google, Google Wallet, μεγάλες αυτές τις εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και ο, ο πελάτης του μέλλοντος δεν ενδιαφέρεται ποιος του δίνει την υπηρεσία που χρειάζεται, αν είναι μια μεγάλη παραδοσιακή τράπεζα ή κάποια μοντέρνα startup. Άρα θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε. Μόνο λοιπόν αν υπάρχουν ίσε ευκαιρίε για, όλα τα, για όλου του φορεί αυτού, θα υπάρξει πραγματική καινοτομία. Και τέλο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πειραματισμού με τη FinTech στην Ευρώπη. Να επιτρέψουμε τον έλεγχο νέων καινοτομιών για να υπάρχει σωστή τεχνογνωσία, εμπειρία, χωρίς να διακυβεύονται τα συμφέροντα του καταναλωτή. Το θέμα δεν είναι να υπάρχουν εξαιρέσει από τον, ε, την νομοθεσία. Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να επικεντρωθούμε στις ευκαιρίες, όχι στα προβλήματα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης σε όλα όσα έχει να μας προσφέρει η FinTech για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε την οικονομική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις εξελίξεις αυτές. Και αυτό επειδή η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε αδύναμη θέση, αλλά όπως και ο Ολλανδός Μαξ από τη Φόρμουλα 1 θα πρέπει να κάνει πολλούς περίπλοκους ε, ελιγμούς για να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό. Είναι σαν το Φστάπαν ε, η Ευρώπη. Εν δυνάμει αθλητήσε παγκόσμιο. Αλλά θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε αλλαγέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και την συγκεντρία, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα να ξεκινήσουμε με του κοιόδη. Πρώτο, είναι ο κύριος Μπράιν Χέις από το Ελεκτρία, Τρία λεπτά Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και η συγγήτρια έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αλλά και οι άλλοι σκιώδεις συγγητές ε, για το σύνολο. Είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εργάζεται πάνω σε μια task force και περιμένουμε μια έκθεση η οποία θα είναι μια πρεμιέρα στον προσδορισμό των προτεραιοτήτων που θέλουμε, ελπίζουμε βέβαια ότι θα υιοθετηθεί, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ρυθμίσουμε. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή ισορροπία μεταξύ και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ώστε ο κανονισμός που με δυσκολία μπορέσαμε να ε, υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε ε, τα τελευταία χρόνια για έναν ασφαλή χρηματοπιστωτικό, μια ασφαλή χρηματοπιστωτική τάξη, θα φέρει καλά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή την καλή ισορροπία. Και πρέπει να πω επίσης, όπως πήγε η συγγήτρια, ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται στην καλύτερη θέση στην υπόθεση αυτή. Αν κοιτάξουμε δηλαδή τις επενδύσεις στον χώρο αυτών τα τελευταία χρόνια, δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα στην Ευρώπη. 22 δισεκατομμύρια επενδύσεων του 2015 σε όλο τον κόσμο, μέχρι 500 εκατομμύρια πέρσι. Ε, παρουσιάζεται λοιπόν μια εκθετική ανάπτυξη και η Ευρώπη πρέπει και να καλύψει το χαμένο έδαφος και να εξασφαλίσει πεδίο για τη χρηματοδότηση και την έρευνα που θα στηρίξει τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτό το νέο καινούριο χώρο. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικά κέντρα που επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτής, αυτού του χώρου που βρίσκεται ακόμη σε εμβριακή κατάσταση. Στη χώρα μου έχουμε ήδη μια καλή ανάπτυξη, πρέπει να γνωριστεί και αυτό. Και η έκθεση όπως και οι τροπολογίες που έχουμε εξετάσει ιδιαίτερη σημασία έχουν γιατί προσδιορίζουν προτεραιότητες και χωρίς να θέλω να επαναλάβω τα όσα είπε η συγγήτρια έχει μεγάλη σημασία η έμφαση στην κυβερνοασφάλεια αλλά ιδιαίτερα ο χώρος για τις ρυθμιστικές αρχές που θα πρέπει να έχουν την ε, ε, γνώση, την τεχνογνωσία, τα σημεία αναφοράς ώστε να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν το πεδίο εκείνο το οποίο θα επιτρέψει στις μικρές, όλες τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Χρειάζεται δηλαδή διαλειτουργικότητα για τις ρυθμιστικές αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει για μας. Και πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το τεράστιο δυναμικό της ε, CMU ως κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων και των επενδύσεων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν μαζί με την ψηφιακή αγορά. Γιατί 200 εκατομμύρια επιχειρήσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση σε χρηματοδοτικές δυνατότητες. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανάπτυξη και της CMU αλλά και της ε, της ΤΠΕ δηλαδή, αλλά και της FinTech. Είναι μια κατάσταση από την οποία μπορούμε όλοι να αποφεληθούμε και οι επιχειρήσεις και βέβαια οι επενδυτές, ας μην είμαστε όμως, ας μην εθελοτυφλούμε, διότι μπορεί να έχει και στρεβλωτικό χαρακτήρα αυτό το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να περιοριστεί στο δυνατόν το κόστος των συναλλαγών και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλώτες αλλά και η χρηματοοικονομική σταθερότητα που πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των επιλογών και των εξελίξεων. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Παρακαλώ. Εκ μέρου του κυρίου Σωρίνη, κυρία Κάιλη. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου του κυρίου Ελλήνων που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Θα σας ε, παρουσιάσω την τοποθέτησή του. Συγχαρητήρια καταρχάς στην εισηγήτρια την Κόρα για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Είχαμε πολύ καλό και επικοδομητικό διάλογο. Δεδομένα λοιπόν τεχνολογία, χρήματα και κεφάλαια είναι το θέμα μας. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναπτυσσόμενες στις αγορές και χώρος επαρκής πιστεύουμε για καινοτόμους νέες ε, παρουσίες. Παρακολουθώντας τόσο τεκταίνοντας στι στις ΗΠΑ και την Ασία, διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει πρωτοπορία ακόμη, γιατί σημαντικά βήματα δεν έχουν αγωμένα ληφθεί και οι κανονισμοί που υπάρχουν πολλέ φορέ δεν έχουν υποστηρίξει την καινοτομία. Προσπαθούμε λοιπόν να εστιαστούμε στα εξή ζητήματα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει ένα σχέδιο δράση FinTech με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικού και ανοιχτού κατά το δυνατό χρηματοπιστωτικού συστήματος με χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία του καταναλωτή. Οι καινοτόμε χρηματοπιστωτικέ χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε πρέπει να είναι διαθέσιμε με τη σύγκληση και με ρυθμιστικέ προσεγγίσει, χωρί όμω αυθαιρεσία προ όφελο των επιχειρήσεων και των ευάλωτων καταναλωτών. Τα νέα μέσα επικοινωνία. Ε, θα πρέπει να είναι στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία. Οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, πλέον οι ψηφιακές ε, δεξιότητες ή ε, ε, καθοδήγηση που θα πρέπει να προσφέρουμε στον καταναλωτή, η οικονομική κατάρτιση, δηλαδή η γνώση της ψηφιακής αλλά και της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την αποσκόπτη λειτουργία της FinTech στην κυβερνοασφάλεια ιδιαίτερα εστιαζόμαστε στην ασφάλεια των δεδομένων, στους κινδύνους από την ε, ψηφιακή τεχνολογία και εδώ θα πρέπει στο πρόγραμμα δράσης FinTech ε, και το σχετικό νομοθετικό πλέγμα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και τον καταναλωτή. Ε, νέες ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής όπου υπάρχουν κενά πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, σε όρους νομοθετικούς και ρυθμιστικούς Ιδιαίτερα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να αποφευχθούν παράνομες δραστηριότητες φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και νομοποίηση παράνομων εσόδων χάρη στον bitcoin, αλλά, coin, αλλά θα πρέπει και να δούμε τα θετικά της τεχνολογίας αυτής. Εν έλλη χρειαζόμαστε ένα γενικό ε, καλό διάλογο μεταξύ DAX, FinTech και ρυθμιστικών αρχών. Για άλλη μια φορά συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Ήταν πολύ καλή και σημαντική αυτή η εκκίνηση και ελπίζουμε ότι θα φέρει καλά αποτελέσματα για τη FinTech στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και για το ECR ο κύριος Φόξ δεν φαίνεται να είναι εδώ. Από την ΚΟΕ τώρα. Παρακαλώ, κύριος Παδημούλης. Thank you, On behalf of Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο όνομα της Μαρία Ματίας που είναι σκιώσης συγητής και που θα φτάσει αργότερα απόψε στις Βρυξέλλες. Θα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αλλά και για τις συμβαστικές λύσεις που μας έστειλε από την αρχή τη συζήτηση για το FinTech η πολιτική μας ομάδα και ο εισηγητής μας έχει εκφράσει τις ανησυχίες της υπάρχει μια μονόπλευρη προσέγγιση και βασιζόμαστε ουσιαστικά ε, στο ότι η προτεραιότητα δίνεται στους, ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τόσο στους υπάρχει έλλειψη ρύθμισης και δεν γίνονται ε, συγκεκριμένες προτάσεις για να καλυφθεί αυτό το κενό. Γενικά είμαστε επικριτικοί απέναντι σε αυτό το πλαίσιο της κεφαλιακής ευρωπαϊκής αγοράς. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Αυτά είναι βασικά στοιχεία της ανάπτυξης του συγκεκριμένου πλαισίου και αυτά λείπουν από την έκθεση αυτή. Δεν συμφωνούμε ότι το Priori Thinknet θα οδηγήσει ε, σε καλύτερη ρύθμιση και σε καλύτερα αποτελέσματα. Βεβαίω προκύπτουν διαφορετικά ρυθμιστικά προβλήματα ανάλογα με την τεχνολογία. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αύξηση τη ταχύτητα των οικονομικών αποφάσεων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώ. Χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση, καλύτερη προστασία δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφέστεροι περιορισμοί και να υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες ε, κανονιστικών πλαισίων. Ε, αυτά λείπουν από την έκθεση. Το, outsourcing εκ νέου 10 χρόνια μετά την οικονομική, κρίση δεν είναι ένα καλό νέο. Η έκθεση αυτή βεβαίως βελτιώθηκε σε ό,τι αφορά την, προστασία του καταναλωτή κάπως ε, στην διαδικασία που ακολουθήθηκε και αυτού το καλωσορίζουμε, αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο να προσθεθούν πολλά περισσότερα στοιχεία έτσι ώστε ο καταναλωτής να νιώσει ότι συμμετέχει ε, με δίκαιο τρόπο και ότι δεν απειλείται από τις νέες τεχνολογίες για τις μεγάλες επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν θα πρέπει αυτή η πτυχή να ενισχυθεί σημαντικά. Η εκπαίδευση, η ενημέρωση του καταναλωτή πρέπει να είναι κύριο μέλημά μα. Γίνονται κάποιε αναφορέ έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση και αυτό είναι θετικό. Τέλο, υπάρχει το θέμα τη ιδιωτική ζωή και τα ζητήματα παρα... τη παρακολούθηση τη προστασία των δεδομένων που θα πρέπει να υπογραμμιστούν περισσότερο. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή την εισηγήτρια μάλλον για το έργο της και βεβαίως θα στείλω τα μηνύματα της συζήτησης της της εισηγητριά μας. Ευχαριστώ για τους πράσινους τώρα, ο κύριος Ρέιμον. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ε, τον ε, εισηγητή για το έργο του. Ήταν πολύ ε, επικοδομητική η δουλειά που έγινε με τους κοιόδους εισηγητές. Έχουμε αναφερθεί βεβαίω στα ωφέλη και στου κινδύνου αυτών των νέων τεχνολογιών στην έκθεση και αυτό είναι καλό, διότι είναι η πρώτη έκθεση για το θέμα αυτό ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Από την άλλη, βέβαια, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Πρόκειται για μια έκθεση. Μιλάμε για τα καλά και τα κακά, αλλά δεν παίρνουμε απόφαση για το πώ θα τα ρυθμίσουμε. Στα επόμενα χρόνια όταν θα το βρούμε μπροστά μας το θέμα αυτό, δεν θα είναι τόσο απλό και εύκολο όλες οι ομάδες μας να συμφωνήσουμε δηλαδή. Σε αυτή τη φάση βέβαια ήταν σημαντικό να τεθούν τα θέματα αυτά, ήταν σημαντικό να αναφερθούν οι ανησυχίε. Το Think Tank είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι καλό ή κακό, είναι όπως ένα σφυρί. Μπορεί να, χτίσεις κάτι με αυτό ή μπορεί να καταστρέψεις κάτι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται αλλά και τους κινδύνους με το FinTech. Είναι τεράστιες δυνατότητες που μας δίνονται για να είναι πιο αποτελεσματικές οι αγορές, για να είναι χαμηλότερο το κόστος συναλλαγών. Εφόσον όμως μπορέσουμε να βρούμε ένα σωστό σημείο ισορροπία στο μέλλον, ε, αυτή η έκθεση είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. I Σας ευχαριστώ και δεν βλέπω συναδέλφους από το EFTD και το EMF είναι εδώ. στη διαδικασία Eye έχουμε την Νίνα Κίλη, η οποία έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Συνάδελφε. Ευχαριστώ και εγώ να ήθελα να ευχαριστώ την κόρα για την έκθεση της. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα αυτό για μας. Δεδομένη και της ανάγκης να αλλάξει ο χρηματοδοτικός κλάδος, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι νομοθεσία και θα υπάρξει να είναι προσαρμοσμένη στις μελλοντικές ανάγκες και θα πρέπει η τεχνολογία FinTech σε κάθε περίπτωση να είναι περιεκτική γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν συγκεκριμένε ε, οικονομικέ γνώσει, γνώσεις, γνώσει. γνώσεις και εδώ ο κόσμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει ένα iPhone και δεν τα καταφέρνει. Πολλές φορές λοιπόν δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Επίσης να τονίσουμε ότι πολλές εταιρείες FinTech έχουν την αντρατούση στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό θα έχει την επίδρασή του και σε ό,τι αφορά το μέλλον και τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκή συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτή την ευρωγνωμοσύνη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Κάτι άλλο που με ανησυχεί για τις, ε, στο πλαίσιο του FinTech τις ε, RoboAdvice, αυτές τις παροχές πληροφοριών ε, από ρομπότ. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει εκβάθρον τον τραπεζικό κλάδο. Και είναι σημαντικό στην έκθεσή σου που αναφέρει σε κόρα να λεφθεί υπόψη και ο κοινωνικό αντίκτυπο του FinTech σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Μπάλτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση από δική μου πλευρά θα ήθελα καταρχάς ε, και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την έκθεση την οποία θεωρώ πάρα πολύ επιτυχημένη. Πιστεύω ότι θα πρέπει επί της αρχής να τοποθετηθούμε και να συζητήσουμε για τέτοια βασικά ζητήματα γιατί στην έκθεση περιλαμβάνονται κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά το θέμα είναι το πώς, με την ταχύτητα των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του FinTech, πώς ως νομοθέτες μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία θα είναι, για το θέμα αυτό, το ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε τακτικά, να σκεφτόμαστε τακτικά το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη επισκόπηση για όλα τα νέα καινοτόμα αυτά στοιχεία για να μπορούμε αντίστοιχα να τη δράσουμε. Και ως εκ τούτου είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με τις προτάσεις που έγιναν, αλλά επί της αρχής για το μέλλον, επειδή ακριβώς αυτός ο κλάδος περιλαμβάνει τόσες πολλές αλλαγές και ακριβώς επειδή όλα αυτά κινούνται με ταχύτητα του φωτός, εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να συζητάμε το πώς στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, πώς θα τα μεταχειριστούμε και πώς θα μπορέσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται να αντιδρούμε στις εκάστοτε αλλαγές. Αυτό θα πρέπει να είναι το καθήκον μας ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο θεωρώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και να ομολογήσω ότι συμφωνώ. Η υπερβάνους. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εδώ. Αν με υποστηρίζει ο κύριος Μπάλς, εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε μια νέα μέθοδο λαμφαλούση εδώ για το fintech ενδιαφέρον. Εν πάση αυτή τη στιγμή το κείμενο αυτό είναι καλό που έχουμε μπροστά μα. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί. Τώρα από εκεί και πέρα το πώ θα προσαρμοστεί η νομοθεσία ε, είναι μια πρόκληση. Εγώ ω εισηγήτρια για την νομοθεσία TRIPS αναγνωρίζω ότι αυτή η νομοθεσία έχει συνταχθεί χωρίς να σκεφτούμε τι θα γίνει όταν αγοράζει κάποιος ένα package product ε, με το iPhone. Δηλαδή κάναμε μια νομοθεσία για τους ε, outsiders. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι οι οικονομικές πληροφορίες είναι οι κατάλληλες, αλλά δεν πρόκειται για μια νομοθεσία όπου έχουμε ε, ενσωματώσει τη λογική του FinTech. Όπως και να έχει όμως ε, υπάρχει κάτι το οποίο απασχολούσε και τους φιλελεύθερους και θα πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο. Το θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι κάτι που συνδέεται με την ανάπτυξη του FinTech. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτού στο κείμενο και αυτό είναι θετικό. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας για τις μελλοντικέ συζητήσεις δεν ξέρω τώρα ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε τελικά. Θα δούμε τι θα μας προτείνει είτε η Κομισιόν, είτε ο Πρόεδρος, είτε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουμε θίξει ιδιαίτερα και το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι, είναι η αλυσίδα ευθύνη και οπότε και οι συνθήκες προστασίας του καταναλωτή. Δηλαδή, διότι κλασικά σήμερα η προστασία του καταναλωτή εξατάται τελικά από το τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, από το διανομέα δηλαδή του προϊόντος. Με το FinTech όλο και πιο συχνά θα έχουμε μηχανισμούς διανομής όπου ο παρασκευαστής του προϊόντος θα έχει άμεση πρόσβαση στον καταναλωτή. Οπότε αυτή η αρχή της αλυσίδας ευθύνης θα διαταραχθεί. Και θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή μας στις μελλοντικέ μα εργασίε, εργασίες, ιδιαίτερα στις εργασίες ε, για τη συνέχεια που θα δοθεί σε ό,τι αφορά την νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα των ε, χρηματοοικονομικών ε, λιανικών υπηρεσιών, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. αυτό που έκανε το Κοινοβούλιο όπου εξετάσαμε την αλυσίδα ε, παρα, ε, ευθύνης ε, σε άλλα νομοθετήματα, αυτά θα πρέπει να το κάνουμε και εδώ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Να επιτρέψουμε την ανάπτυξη του FinTech, αλλά να προασπίσουμε την αρχή της προστασίας του καταναλωτή. Μάλιστα, ευχαριστώ. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που σχετίζονται με αυτό που είπατε στον φάκελο για το PST. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. βεβαίω, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Η έκθεση είναι ισορροπημένη. Και ε, τα, η τροποπολογία συμβιβασμού. Το FinTech ε, προσπαθεί να πετύχει μια σειρά από στόχους που ορισμένες φορές ε, είναι καταγωνιστικοί μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε ισορροπημένα. Όπως είπαν πολλοί ομιλητές, εδώ δημιουργούνται τεράστιες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και για την πρόσβαση σε άλλες αγορές για τους παρόχους αυτούς. Επίσης ε, αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα του χρηματοοικονομικού κλάδου και οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό διότι θα ανοίξει και στου περισσότερου παίχτε η αγορά. Αυτά είναι θετικά, αλλά από την άλλη θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σαφή πολιτική, ένα σαφές πλαίσιο για τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι κρίσιμος παράγοντας για το FinTech. Ακαιρεότητα λοιπόν και ασφάλεια των δεδομένων αυτών σε μια πολιτική η οποία θα είναι τεχνολογικά ουδέτερη και που θα βασίζεται και στην αρχή της αναλογικότητας. Η προσέγγιση μας βασίζεται στον κίνδυνο, εξετάζουμε δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό κινδύνου για να δούμε ποιοι κανόνες θα εφαρμόζονται. Αναμένουμε με ανυπομονησία την τελική έκθεση. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα και δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Ιουνίου και από εκεί πέρα η Κομισιόν θα αποφασίσει ποιες πρωτοβουλίες ε, θα πάρει, ποια μέτρα θα προτείνει και θα υποβάλει μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και όλους αλλά και τους λοιπούς ομιλητές για την υποστήριξη είναι σημαντικό το ότι διατυπώσαμε εδώ κάποιες κοινέ αρχές. Δεν έχουμε βέβαια απαντήσει σε όλα τα προβλήματα, δεν είναι πανάκια αυτό το κείμενο, αλλά θέτει τα σωστά ερωτήματα. Αυτό το κάναμε. Πιστεύω, πολλοί από εσά ε, ε, αναφέρθηκαν στην ανάγκη ε, ταχύτητας, υπερβώς αναφέρθηκε σε συστήματα ε, αξιοπιστίας, η ΓΚΟΕ αναφέρθηκε στο σωστό σημείο ισορροπία σε σχέση με τα συμφέροντα και των καταναλωτών, σε σχέση μεταξύ συμφέροντων καταναλωτών και εμπορικών συμφερόντων. Ε, θα πρέπει βεβαίω να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία. Οι συστάσει μα πάντω από το Κοινοβούλιο μπορούν να αποτελέσουν μια καλή συνεισφορά εν ώψη του σχεδίου δράση FinTech τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι ένα πραγματικό σχέδιο δράση με συγκεκριμένε δράσει και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διότι μόνο δύο επιλογές έχουμε σε ό,τι αφορά το μέλλον της FinTech. Είτε ε, κάποιος κάθε στο τραπέζι, είτε αποτελεί μέρος του μενού για να τον φάνε. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αύριο θα λάβει χώρα ψηφοφορία και 31 Μαΐου στην Ολομέλεια. Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο, μάλλον στο προηγούμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, τη γνωμοδότηση σε σχέση με τις πολιτικές ελάχιστου εισοδήματο για την αντιπολέμηση τη φτώχειας. Ο κύριος Ριέγας είναι ο εισηγητής και έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευελιξία που μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ σήμερα παρά την καθυστέρηση της πτήσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους μου το επιτρέψατε αυτό. Θα προσπαθήσω να μην σας καθυστερήσω. Έχετε ένα αντίγραφο του σχέδιου γνωμοδότησης. Ε, είναι σαφής η γνωμοδότηση, είναι απλή είναι σύντομη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, σε αυτό το πρώτο σχέδιο κειμένου, είναι να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση ρεαλιστική. Πρώτα απ' όλα. Μια προσέγγιση με βάση αντικειμενικά στοιχεία. Η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Η κοινωνία δεν είναι τέλεια. η οικονομία της αγοράς έχει επιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να αποφύγουμε και τα κράτη πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους για αυτές τις επιπτώσεις. Τα στοιχεία αυτά ε, δεν είναι δικά μου και αποτυπώνουν την φτώχεια και το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι ε, ζουν σε συνθήκες φτώχειας πολλοί διεθνείς φορείς έχουν αναφερθεί στη σημασία των δημοσίων πολιτικών των πολιτικών αναδιανομής χωρίς τις οποίες τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Και βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας που ήρθαν να επιδεινώσουν αυτούς τους δείκτες. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία. Δεν νομίζω να μπορεί κανείς να τα στρεβλώσει ή να τα αμφισβητήσει. Και αυτή είναι και η βάση της έκκλησης που απευθύνουμε. Ελπίζουμε ε, η επιτροπή αυτή να την ασπαστεί. Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την οικονομική πραγματικότητα που ζουν οι συμπολίτες μας ε, το οικονομικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, που έχει οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις στο να έχουν μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική, όλα αυτά μας οδηγούν σε μια πραγματικότητα ε, που μας υποχρεώνει ε, να χαράξουμε πολιτικές οι οποίες να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα, διότι αν το δούμε αυτό ως μέρος των μακροοικονομικών δικτών που χρησιμοποιούμε, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το ΑΕΠ και για κάποιους ε, αμυγός οικονομικούς δείκτες. Θα πρέπει να υπάρχουν οι δείκτες και για την ανισότητα στην κατανομή των εισοδημάτων. Θα πρέπει να προσέξουμε τους θύλακες φτώχειας που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Μιλάμε εδώ λοιπόν για δημόσιους πόρους που δεν διατεθέτουν τα κράτη-μέλη λόγω δημοσιονομικών περιορισμών και που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί το θέμα της στόχιας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος. Αυτό δεν είναι μια ιδέα της ΓΚΟΕ. Είναι μια ιδέα των μεγάλων διεθνών οργανισμών. Αυτοί ζητούν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. και η αναφορά, ε, μάλλον το, το ύψος αυτού του εισοδήματος, σύμφωνα με τις οργανισμούς, πρέπει να είναι 60% του μέσου μισθού, του μέσου εισοδήματος. Αυτό είναι, αυτή είναι η καρδιά της πρότασής μας. Θα τα βρείτε τα υπόλοιπα στο κείμενο. Είμαστε ερεθιμένοι να δεχθούμε οποιαδήποτε συνεισφορά έρχεται να βελτιώσει αυτό το κείμενο και θα εργαστούμε συνενετικά έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα όσο γίνεται πιο ευρύ συμβιβασμό. Για το ΕΛΚ, η κυρία Μαλέτιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα παρουσιάσω το σημείο που α, έχει προετοιμάσει η σκέψη μας, η κυρία Ραμαντώντς. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μικέλ Βιέγκας για τη δουλειά που έχει κάνει. Και τα τρία βασικά σημεία τα οποία έχει προετοιμάσει η κυρία Ρωμάνα Τόνς είναι τα εξή. Πρώτον, τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προσωρινά χρηματοοικονομικές ε, δυσκολίες. Αλλά εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να τα αναπτύξουν αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Όλοι ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό είναι να δίνετε ευκαιρίες στον κόσμο να φροντίσουν τις οικογένειές τους και τους εαυτούς τους, δίνοντας κάποια ελάχιστα βιωτικά επίπεδα και να μην υπάρχει εξάρτηση. Ελάχιστη ελάχιστο εισόδημα, το κατώτατος μισθός βοηθά. Βοηθά αυτούς που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν ρυθμίζει το θέμα της ένδυας, της φτώχειας. Δεν λύνεται έτσι το θέμα της φτώχειας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεύτερο σημείο. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική δομή, διαφορετική οικονομική ισχύ και με, έχουν διαφορετικές ικανότητες για να παρέχουν πόρους. Να μην ξεχνάμε ότι η παροχή ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί μια υποχρέωση η οποία βαρύνει οικονομικά τα κρατημέλη. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να κινηθούμε πιο πολύ προς την κατεύθυνση του να δίνουμε κίνητρα στην οικονομία και να δημιουργούμε καινούριες θέσεις εργασίας για να υπάρχει ανεξαρτησία, χωρίς οικονομική εξάρτηση. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Τρίτο σημείο τώρα της συναδέλφου, η σύνδεση της χρηματοοικονομικής ε, πειθαρχίας δεν αποτελεί σωστή βάση για τις συζητήσεις μας. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα εξασφαλίσουμε σωστό τρόπο δαπανών αποτελεσματικές επενδύσεις και αποτελεσματικές δαπάνες των δημοσίων πόρων. Και αυτό θα πρέπει να διέπει όλες τις συζητήσεις για τα κοινωνικά δίκτυα και τις δικλείδες κοινωνικής ασφάλειας και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες. Άρα, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Η κυρία Περές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Μουρέλα, ο οποίος ε, λείπηκε. Λόγω δραστηριοτήτων που τον ε, απασχολούν. Ε, χαίρεται ιδιαίτερα για την ε, μελέτη του θέματος ενλώσεων ελέγχου του εισοδήματος ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. βέβαια και μέσω των εκλογικών διαδικασιών μπαίνει το θέμα αυτό θεωρεί ότι πρέπει να συνδυάζεται η ευπευθυνότητα και η αλληλεγγύη ιδιαίτερη έμφαση εκδοθεί μέχρι τώρα από ό,τι σημειώνει στην ευθύνη με αιμονή στις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κατά τρόπο όμως και τυφλό πολλές φορές κοινωνικά. Ιδιαίτερα λοιπόν ενδιαφέρεται για τις ε, επιλογές της Επιτροπής Απασχόλησης και τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές ε, πολιτικές, νομισματικές πολιτικές μπορούν να ε, οδηγήσουν σε κοινωνικές αλλαγές. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί την γνωμοδότηση αυτή. Θέλει να χαιρετήσει τι προσπάθειες του εισηγητή για και τη δουλειά του και συμμερίζεται την πεποίθησή του ότι θα πρέπει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η γνωμοδότηση να παραμένει ορατό. 24% σημειώνει του πληθυσμού βρισκόταν ε, σε επίπεδα φτώχειας και αποκλεισμού. Για το ημείωση λοιπόν των ανισοτήτων, ιδιαίτερη σημασία έχει και η απώλεια περιουσίας αλλά και η απώλεια εισοδημάτων. Στόχοι λοιπόν μια στρατηγικής 2020 καλώς νοουμένη και θεωρεί ο ισχυώδης ότι θα πρέπει να ε, εισαχθούν σωστοί δείκτε μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, δεσμευτικοί μάλιστα, ώστε τα μέτρα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και τις ανισότητες αλλά και το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης για το οποίο οφείλουμε να διαπιστώσουμε πως αναπτύσσεται πολύ πιο βραδέως από ότι ο πληθωρισμός και άρα οδηγεί σε ανισορροπία σοβαρή. Τροπολογίες θα καταθέσει από ό,τι διαπιστώνουμε στο πνεύμα αυτό. Θεωρεί ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει οδηγία πλαίσιο για ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα. Επίσης θέλει να ε, σημειώσει ότι το Διεθνές Ταμείο έχει τον τρόπο να επηρεάσει τους πολλαπλασιαστές, τους οικονομικούς πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιεί η Ένωση και αυτό σημαίνει πολιτικές εσόδων. Και αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν ότι οι πολιτικές των εσόδων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημοσιονομική ανάπτυξη προς την ανάπτυξη την οικονομική και τη μείωση των ανισοτήτων. Σημειώνει επίσης ότι οι χώρες όπου υπάρχει ένα στεναρό σύστημα ελάχιστου εισοδήματο έχουν μπορέσει να ξεπεράσουν με λιγότερη επιδείνωση, μικρότερη επιδείνωση των ισοτήτων την κρίση και αυτό βέβαια αντικατοπτρίζεται και στην θέσπιση των αυτόματων σταθεροποιητών. Προσωπική τώρα παρατήρηση, η Επιτροπή στην προηγούμενη της ε, σύνθεση είχε διατυπώσει τέτοιου είδου συστάσει. Κάτι ακόμη που θέλει να σημειώσει ο συνάδελφος είναι ότι στο θέμα του ελάχιστου οικουμενικού ελάχιστου εισοδήματο. Με συγχωρείτε λέει ο μιλήτρια, χάσα τα λόγια μου. Το θέμα λοιπόν του ελάχιστου ή βασικού οικουμενικού εισοδήματο έχει ήδη καλυφθεί από μια πρωτοβουλία πολιτών το 2013, ότι έχουν γίνει παραδείγματι εργασίες στο πλαίσιο της γαλλικής γερουσίας και ότι ήδη αναπτύσσεται σχετική ε, απόπειρα και δοκιμαστική εισαγωγή στη Φιλανδία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει και δημόσια διαβούλευση αλλά και να εξετάσει όλε τι δυνατότητε για το θέμα αυτό. Σημειώνει επίση ότι το θέμα τη οικονομική αλληλεγγύη και τη αντιμετώπιση των ανισοτήτων έχει ουσιώδη σημασία σε χρονική στιγμή όπου ορισμένε εκλογικέ αναμετρήσει δείχνουν ότι η Ευρώπη θεωρείται πω επιδεινώνει τι ανισότητε και αυτό απειλεί ήδη το μέλλον και την επιβίωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. και αν μου επιτρέπετε πρόεδρε μια προσωπική ακόμη παρατηρήση για ένα-δύο λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω ότι πέραν των ε, εργασιών που έχουν ήδη ε, αναπτυχθεί η έκθεση Φιγκεϊρέιδου παραδείγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σταθεροποιητικό ρόλο ενό ελάχιστου εισοδήματο, όπω είχε σε μια μελέτη της το θέμα του ελάχιστου μισθού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί εδώ γίνεται πολύ συχνά αναφορά σε έναν μέσο μισθό. Ωστόσο, δεδομένης της κατολίστησης των μισθών σε ορισμένα πρέπει να κάνουμε αναφορά μάλλον σε όριο φτώχειας. Και αυτό θα ήταν πολύ πιο σωστή επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Το ECR με τον κύριο Λούκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση για την οποία όμως θεωρώ ότι θα έπρεπε να ήταν λιγότερο γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ και περισσότερο της ΓΚΟΕ ως ομάδας. Θα χρειαστεί πολύ ακόμη δουλειά για να εξασφαλίσει πλειοψηφία αυτή η πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα συνιστούσα να γίνεται διαφοροποίηση ως προς τις έννοιες φτώχεια και ανισότητα. Η ανισότητα είναι μια έννοια πολύ δύσκολο να περιγραφεί και ποσοτικά πάνω απ' όλα να προσδοριστεί, αλλά είναι και δύσκολο να προσδιοριστούν μέτρα του τι σημαίνει ανισότητα μέσα σε ένα κράτος, μέσα σε μια κοινωνία. Δεδομένου ότι η ισότητα είναι μια αξία προς την οποία πρέπει να τίνουμε, θα μπορούσαμε να μιλούμε για, μια πιο αποτελεσματική, για ένα πιο αποτελεσματικό καταμερισμό της εργασίας, της οικονομικής δραστηριότητας και βέβαια αναλόγως εισοδημάτων. Άρα λοιπόν πρέπει περισσότερο να επιμείνουμε στην ε, ισότητα, στην έννοια τη ισότητα μέσα αυτή την νομοδότηση, η οποία είναι σύντομη πολύ και δεν θα μπορούσε να έχει πολύ περιπλοκέ έννοιε. Η φτώχεια επίση είναι μια διαφορετική έννοια. Στον προσδιορισμό λοιπόν της φτώχειας, εγώ θα έτεινα να προτείνω μια απόλυτη, έναν απόλυτο ορισμό και όχι σχετικό, όπως 60% επί του μέσου εισοδήματος που αναφέρεται εδώ, γιατί αυτό μπορεί να ορίσει ένα ελάχιστο επίπεδο φτώχειας ανεξαρτός του πλούτου μιας συγκεκριμένη κοινωνίας. Ανεξάρτητη λοιπόν η φτώχεια από το επίπεδο πλούτου μιας κοινωνίας. Στο ελάχιστο εισόδημα τώρα. Μου φαίνεται καλή αυτή η έννοια, αλλά βέβαια πρέπει να συζητήσουμε το ύψος αυτού του ελάχιστου εισοδήματος εξασ είναι ε, βέβαια δεδομένο ότι χρειάζεται να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο εισόδημα, αλλά πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με ένα ελάχιστο μισθό. Το ελάχιστο εισόδημα σημαίνει ότι εάν το δεχθούμε δεν μπορούμε να έχουμε και την έννοια του ελάχιστου μισθού ταυτόχρονα. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προτιμηθεί η έννοια του ελάχιστου εισοδήματος σε σχέση με αυτήν του ελάχιστου μισθού. Αυτό που δεν βλέπω όμως στην προσέγγιση στην γνωμοδότηση, για να το πω διαφορετικά, αυτό που θα ήθελα στην ε, γνωμοδότηση αυτή να τονιστεί λιγότερο, είναι η έννοια της αναδιανομής. Εδώ η φτώχεια παρουσιάζεται ως ένα ε, φαινόμενο το οποίο μπορεί με την αναδιανομή του πλούτου να αντιμετωπιστεί. Ενώ εγώ θεωρώ ότι πρέπει με την ανάπτυξη να επιδιώξουμε πρόσθετα εισοδήματα, άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες, ε, δυνατότητε για ανάπτυξη μεγαλύτερου εισοδήματο και όχι αναδιανομή. Η έννοια λοιπόν της οικονομική ανάπτυξη για μένα χρειάζεται να ενισχυθεί περισσότερο μέσα σε ε, αγορές εργασίας που θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση της νομοδότης. Τον μιλούμε για στήριξη του εισοδήματος, τον μιλούμε για κλιμάκωση των μισθών, ε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τονίσουμε την έννοια αυτή με εισόδημα το οποίο δεν θα εξαρτάται από την εργασία, που δεν θα προκύπτει από την εργασία. Μια επικοδομητική βεβαίως προσέγγιση θα είναι να μην εξασφαλίσετε ένα εισόδημα μόνο με υπερβολική χρέωση, αλλά περισσότερο θα πρέπει να προσφεύγουμε στις επενδύσεις. Η σταθερότητα φορολογική έχει πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως και πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία ε, πλήττονται από υπερβολικό Χρέο Και πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σημειώνω δε ότι δεν μίλησα τόσο όσο η κυρία Μπέρε. Σα ευχαριστώ. Και δεν βλέπω κανέναν από την ομάδα των φιλελευθερών. Ο κύριο Ούρθασον από τους πράσινου, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βέιγας για την παρουσίασή του ε, και για το έργο του. Είναι μια πολύ καλή βάση το κείμενο για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ καιρό. Πριν από μερικά χρόνια υπήρξε μια έκθεση της, ΕΟΚΕ ε, για ένα ελάχιστο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να το ξαναδούμε μάλιστα, να ξαναδούμε αυτή την έκθεση, διότι περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε, το είπε και η κυρία ε, ότι πρέπει να βρούμε μηχανισμού βάσει των οποίων όχι μόνο θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ανισότητα, αλλά θα πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, παίρνονται μέτρα συνοδευτικά, ε, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι ε, η αρχή πτέρνα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να γίνει κατανοητή και να τύχει υποστήριξη από τον πληθυσμό αυτά που αναφέρει η γνωμοδότηση λοιπόν είναι σωστά. Υπάρχει και ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να το πούμε εμείς ως ΕΚΟΝ. Βεβαίως υπάρχει ένας οικονομικός αντίκτυπος, εξαιρετικά σημαντικός, ε, λόγω αυτών των θυλάκων φτώχειας. Σε, κάποιες, σε κάποια κρατημέλη Έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ανεργία και αυτοί οι θύλακε φτώχεια ε, έρχονται ε, να φρενάρουν, να σταματήσουν τους ρυθμού ανάπτυξη. Το δείχνει αυτό, το δείχνουν και εκθέσει του ΩΣΑ μεταξύ άλλων. Ε, είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα του ρυθμού ανάπτυξη. Βεβαίω και συνδέεται με την ανισότητα αυτό. Αφορά τη φτώχεια, αφορά και την ανισότητα. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να ασχολείται και με τα δύο η έκθεση. Το Δούνο του ε, λέει στην έκθεσή του ότι εφόσον 20% των υψότερων εισοδημάτων συσσωρεύει 1% παραπάνω, ε, έχουμε μείωση του ΑΕΠ 0,08%. Όταν όμως αυτό το 1% πλούτου προσθεθεί στο 20% των πλέον φτωχών, τότε το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,38%. Αυτό τα λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του και μπορώ να τα, μοιρασ... να τα μοιραστώ με τους αδέλφους. Εκεί υπάρχουν κάποιοι συντελεστές εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Ε, και σίγουρα θα υπήρχαν, θα υπήρχαν θετικές επιπτώσεις ε, για την ευρωπαϊκή οικονομία ε, εφόσον είχαμε αυτά τα, αυτό το κειμένο εισόδημα. Να ευχαριστήσω λοιπόν για την φορά του εισηγητή. Ε, θα θέσουμε κάποια ζητήματα βεβαίως ε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να εξετάσουμε μηχανισμούς ελάχιστων ε, εισοδημάτων που υπάρχουν ήδη σε κάποιες χώρες όπως τη Φιλανδία αλλά και κάποιες τοπικές αρχές ε, περιφερειακές ε, ε, σχεδιάζουν παρεμφερή συστήματα από τα οποία θα πρέπει να εμπνευστούμε ε, και να τα αναλύσουμε και βεβαίως η πρόταση μιας οδηγίας προς την κατεύθυνση αυτή μια οδηγία, πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετική. Είμαστε λοιπόν στη διαθεσία για να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Σημείωσα όλες τις προτάσεις που ακούστηκαν, αλλά και τις κριτικές. Ε, όλα αυτά είναι εύστοχα. Βεβαίως εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο κειμένου, έτσι. Το οποίο μπορεί κάλλιστα να τροποποιηθεί. Και βεβαίως είναι ατελές. Είμαι λοιπόν ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση. Και θέλω να εξασφαλίσω ότι αυτή θα είναι ε, μία γνωμοδότηση του συνόλου της ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ και όχι μια ομάδα μόνο. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Θα πρέπει βεβαίως ε, να εργαστούμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα κείμενο Θέλω να τονίσω το εξής. Όπως είπα πριν από λίγο, θα πρέπει να εργαστούμε με βάση πραγματικά στοιχεία, αντικειμενικά. Εδώ, σε αυτό το φαινόμενο, η αγορά έχει αποτύχει. Η αγορά μάλιστα παράγει αυτό το φαινόμενο φτώχειας και θυλάκων φτώχειας. Όταν έχουμε 23% κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτό είναι ανησυχητικό και χρήζει απάντησης. Εάν δούμε ευρύτερα ζητήματα στη συζήτηση αυτή, αν εξετάσουμε κατά πόσο να παρθούν κάποια μέτρα σε επίπεδο προσφοράς, ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε ε, μια πολύ γενναιόδορη πολιτική, ε, ποια είναι τα καλά της, ποια είναι τα κακά της. Ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσουμε σε συμφωνία αν το διευρύνουμε τελικά στο επίπεδο της προσφοράς το ζήτημα και των κινήτρων. Εδώ εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πούμε ότι εκεί όπου υπάρχει, όπου έχει αποτύχει αγορά, εκεί όπου υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά σοκάρει πολλούς συμπολίτε μας ε, τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε. Βεβαίως συμφωνώ ότι εδώ τα κράτη-μέλη έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια κεντρική προσέγγιση σε κεντρικό επίπεδο. Παρ' αυτά μπορούμε με κάποιες ελευθερές γραμμές να πούμε ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου απέναντι στην πραγματικότητα, η οποία ε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους ε, πολίτες της Ευρώπης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έχει κάποιες προτάσεις να κάνει για την αντιμετωπίσή του. Η φτώχεια και η ανισότητα και συμφωνώ, ε, συμφωνώ με κάποια πράγματα που λέξαν ε, για το διαχωρισμό των δύο, αλλά και η ανισότητα έχει τη σημασία της βεβαίως. Δεν μιλάμε εδώ για κάποια χώρα της υποσαχάριας Αφρικής. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα που αφορά την καρδιά της Ευρώπης. Τι μας λέει λοιπόν η ανισότητα αυτή. Μας λέει ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από κάποιες αιτίε. Και αυτό οδηγεί στο να μην γίνεται δίκαια, δίκαια η κατανομή του πλούτου. Ε, στην ίδια περιφέρεια ή στην ίδια χώρα ή στην ίδια ήπειρο υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις στα εισοδήματα. Και αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί με αμυγός με οικονομικούς όρους. δεν είναι απαραίτητη, απαραίτητο να υπάρχει αυτή η ανισότητα. Σα ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα και αναμένω να συνεργαστούμε στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα. Λοιπόν, τροπολογίες ως 4 Μαου. 29 Μαου εξετάζονται τα, οι, οι 8 Ιουνίου στην ΕΚΟΝ. 22 Ιουνίου και τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Πέρας τη συνεδρίαση, αύριο ξεκινούμε 9.30 με την ακρόαση.